εξωτερικής ε, προσέγγισης του ευρώ θα λάβει χώρα αμέσω μετά τη συζήτηση της έκθεσης Λάινεν Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντοοικονομική Λογαριασμή. Μία μικρή τροποποίηση λοιπόν στη μέρησια διάταξη ε, μετά από την οποία μπορούμε να εγκρίνουμε την ε, ημερήσια διάταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, σύμφωνα με τη ημερήσια διάταξη λοιπόν έχουμε το πρώτο σημείο μας αφορά δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω της επαιτίου των μαζικών εκτοπίσεων του 1941 στα κράτη της Βαλτικής. Μετά από την δήλωση θα ακολουθήσει σύντομος γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες οι οποίες ε, θα μιλήσουν για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι γιορτάζουμε την 70η επέτειο των μαζικών εκτοπίσεων στις χώρες της Βαλτικής για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Σοβιετική Ένωση. Έγιναν αυτές οι εκτοπίσεις το 1941 στην περιοχή της Βαλτικής με στόχο να εκτοπιστεί ο πληθυσμός της Εστονίας, Λιθουανίας και Λετωνίας και επομένως να εξαλειφθούν οι κοινωνικές και πολιτικές ελίτ της χώρας των χωρών αυτών. Πρόκειται για επιστήμονες, για πολιτικούς, πρόκειται όμως και για άτομα τα οποία έδειχναν μια ανεξάρτησία σκέψης. Πρέπει να σκεφτούμε τις ε, δεκάδες χιλιάδες θυμάτων της τρομοκρατίας από τη Σοβιετική Ένωση εκείνη τη χρονική στιγμή. Όλα αυτά μας ενδιαφέρουν όλους μας. Όλους μας. Πρέπει να σκεφτούμε όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν κατά του ολοκληρωτικού συστήματος στη Σοβιετική Ένωση, το οποίο κατέστηλε τις ελευθερίες των λαών. Τα βάσανα αυτών των λαών τους έδωσαν και τη δύναμη ώστε μετά από 50 χρόνια να μπορέσουν να επανέλθουν στην Ενωμένη Ευρώπη. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στις 22 Ιουνίου, σε δύο εβδομάδες περίπου, θα γιορτάσουμε και την ευδικο, ευδικο, ευδομικοστή επέτειο της ε, επίθεση της Γερμανίας κατά της Σοβιετικής Ένωσης που ήταν και το τέλος του συμφώνου ε, Μολότοφ-Ρίμπεντροπ και επομένως είναι μια σημαντική επέτειο στην οποία θα πρέπει να ενθυμηθούμε για την ιστορία την ευρωπαϊκή. Σκεφτόμαστε ιδιαίτερα τους συναδέρφους μας από την Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία η μοίρα των χωρών αυτών όμως μας κατέδειξε ότι η Ευρώπη μπόρεσε να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες και τις εσωτερικές εντάσεις. Για τον λόγο αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία των συναδέλφων μας από τις χώρες αυτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ενθυμούμαστε αυτό στη σημερινή ημέρα. Περνάμε τώρα στις ε, παρεμβάσεις από τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Τούνε Κέλαμ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από 70 χρόνια, περίπου 50.000 Λιθουανοί, Λετονοί και Εστονοί εκτοπίστηκαν με δύο τρόπο από τις στίες τους στα βαλτικά κράτη τα οποία ήταν υπό την Σοβιετική κατοχή. Αν συγκρίνουμε αυτό τον αριθμό, τις 50.000 με τον πληθυσμό που ήταν τότε 5,5 εκατομμύρια των τριών αυτών χωρών, αν δούμε τι θα σήμαινε αυτό για μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, θα είχαμε κάτι της τάξης των 430.000 πολιτών από το Ηνωμένο Βασίλειο ή 363.000 από την Γαλλία. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι αντίστοιχο στο Ηνωμένο Βασίλειο ούτε στη Γαλλία. Το Μάιο του 1941 η Σοβιετική ηγεσία αποφάσισε να υπάρξει αυτή η εκαθάριση των αντισοβιετικών στοιχείων στην Λετωνία, Λιθουανία και Εστονία. Όπως είπε και ο Πρόεδρος μας, ήταν η εκαθάριση των πολιτικών και οικονομικών και πνευματικών ελίτ. Τα άτομα αυτά εκτοπίστηκαν στην Σιβηρία και στο ναρκτικό κύκλο για να αντιμετωπίσουν πείνα και βάσανα πολλοί πήγαν σε στατόπεδα συγκέντρωσης χωριστά από τις οικογένειές τους όπου έχασαν τη ζωή τους. Σε πολλές ε, περιοχές περίπου 50% των, ε, ε, των εκτοπισμένων έχασαν τη ζωή τους. Ήταν ένα μεγάλο πλήγμα στη δημοκρατική κοινωνία των πολιτών στις χώρες της Βαλτικής. Αυτές οι αδιάκτητες εκτοπίσεις οδήγησαν σε βαθιά ψυχολογικά τραύματα για τα θύματα που ζήσανε επί πολλά χρόνια κάτω από τέτοιες συνθήκες και αυτό τους οδήγησε να αποδεχθούν και την καταστολή και την λογοκρισία, τους έκανε να πιστεύουν ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει δημοκρατία εκεί. Ο Σέργεϊ Κοβαλιόφ, το βραβείο Σαχάριοφ, Σαχάροφ, τόνισε ότι με τη σύγχρονη ορολογία επρόκειτο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η ανάμνηση λοιπόν των 70 χρόνων από τις εκτοπίσεις στη Βαλτική είναι και μια ευκαιρία να έχουμε καλύτερη κατανόηση ότι το παρελθόν των λαών αυτών της Βαλτικής είναι και το παρελθόν όλων των λαών της Ευρώπης. Η ενθύμηση λοιπόν αυτών των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας του 1941 θα πρέπει να είναι κομμάτι αναπόσπαστο της κοινή μας ευρωπαϊκής ιστορίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξή σας και την αλληλεγγύη σας και για το γεγονός ότι τα κράτη των Βαλτικών χωρών έχουν καταφέρει με αυτή την αλληλεγγύη να είναι πλέον κομμάτι της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Ε, Ο κύριος Σφόμποντα έχει το λόγο από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Κέλαμ, αγαπητοί συνάδελφοι από τις Βαλτικές χώρες, αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια στιγμή που πρέπει να ενθυμηθούμε όλοι τη μαζική εκτόπιση των πολιτών ε, των Βαλτικών χωρών. Είναι μια από τις πιο ζωφερές και σκοτεινές στιγμές στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μπορεί επομένως να δικαιολογήσει κανείς ότι από ονομάστηκαν οι εκτοπίσεις του αιώνα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει για το σημείο αυτό μια πλήρης ε, διαλεύκανση της ιστορίας Σοβιετικής Ένωσης και του Σταλινισμού. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει παρά μόνο μία υποστήριξη από όλους για να υπάρξει αυτή η διαλεύκανση της ιστορίας της Σοβιετικής Ένωσης που ακόμα επιρρύπτει σκιές στην ιστορία όλων των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σκεφτούμε όμως και τα θύματα άλλων τέτοιων εκτοπίσεων όπως είναι οι Αρμένοι στην Οθωμανική ε, Αυτοκρατορία την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης και άλλες μαζικές μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που έγιναν λόγω του ναζιστικού και του κομμουνιστικού καθεστώτος. Και μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακολούθησαν μαζικές μετακινήσεις και εκτοπίσεις που άφησαν βαθιές πληγές όπως παραδείγματος χάρη στην ε, πρώην Ιουκοσλαβία. Και επίσης και τα απικιακά καθεστώτα έκαναν αντίστοιχες ε, ενέργειες. Θα πρέπει εμείς λοιπόν να απορρίψουμε όλες αυτές τις δικαιολογίες και τα προσχήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για αυτές τις εκτυπώσεις και να αποδώσουμε δικαιοσύνη όταν αυτό είναι ακόμα δυνατό, όπως τώρα στην περίπτωση του Μπλάντιτς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει τώρα συμπεριλάβει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις ανεξάρτητες βαλτικές χώρες και ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι μιας διαδικασίας που δεν έχει ακόμα τελειώσει, της διαδικασίας της επανένωσης της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε όχι μόνο τους εαυτούς μας, αλλά και αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον εκτοπισμό και τα βάσανα αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δηλώσεις που έχουν γίνει από αυτή την πλευρά οι κοινέ δηλώσεις του Πρόεδρου της Γερμανικής Μπούντεστα και της Πολωνικής Δίαιτας για τις εκτοπίσεις αυτές. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι ένας τρόπος να μας κάνει να σκεφτούμε καλύτερα, να σκεφτούμε τι συμβαίνει με αντίστοιχες αντίστοιχα γεγονότα, όπως τα γεγονότα των, της Αραβικής Άνοιξης και των ατόμων τα οποία εκδιώκονται από τις χώρες τους και έρχονται στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε τη σημασία του εθνικισμού και τις ε, πληγές που προέκυψαν από τους εθνικισμούς στην Ευρώπη, αυτά θα πρέπει να μας ε, οδηγήσουν να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποτρέψουμε γεγονότα τα οποία έριξαν την Ευρώπη σε βαθύ σκοτάδι. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε όλα αυτά τα γεγονότα, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε όλα αυτά τα οποία υπέφεραν οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να καταληφθούμε από την αδιαφορία και θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια νέα Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα ο Λεωνίδας Δόνσκι εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Σας ευχαριστώ. Οι εκτοπίσεις του πληθυσμού των Βαλτικών χωρών το 1941 ήταν από τα πιο δραματικά γεγονότα του 20ου αιώνα η Λετωνία, η Εσθονία και η Λιθουανία έχασαν όλοι τους τη δημοκρατική και πολιτισμένη θα έλεγα ζωή και έμειναν σε απομόνωση για μισό αιώνα. Και έτσι καταστράφηκε και η ενότητα της Ευρώπης. Η απομόνωση αυτή έλξε μόνο το 90. Οπότε και ξαναρχίσαμε να μπορούμε να μιλούμε για αλλαγή στην ιστορία των βαλτικών χωρών. Το 2004, δε, όταν μπήκε στην Ένω, μπήκαν στην Ένωση οι χώρες αυτές, μπορέσαμε να κάνουμε και ένα μνημείο. Οι πιο προοδευτικοί εκπρόσωποι των χωρών αυτών εκτοπίστηκαν. Έτσι ώστε... Και αυτό ήταν μάλλον ένα, μια από τις πιο χαρακτηριστικές πράξεις του σταλινισμού. Ο Στάλιν συνήθιζε να αποκεφαλίζει τις ελίτ των χωρών, των δορυφόρων χωρών. Σήμερα που είμαστε σε θέση να γιορτάσουμε αυτή την 70η επέτειο των εκτοπίσεων, είναι κάτι το σημαντικό γιατί έτσι επανέρχεται η αξιοπρέπεια και η πολιτική μνήμη στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. ο κύριος Ρόμπερτ Ζιλέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά το ότι η εκτόπιση των κατοίκων των βαλτικών χωρών τον Ιούνιο του 1941 και στις 25 Μαρτίου του 1949 ήταν ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα για τους πληθυσμούς των χωρών αυτών Παρόλα αυτά η κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη δεν γνωρίζει ακόμη τα γεγονότα αυτά επαρκώς. Το χιτλερικό καθεστώς έχει καταδικαστεί, αλλά το σταλινικό, η γενοκτονία των χωρών αυτών από τον Στάλιν δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί από όλους. Πολλοί δεν θέλουν καν να το αναφέρουν. Αυτό έχει πολύ αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία των λαών της Βαλτικής. Όπως είπε ο Σολζενίτσιν, υπονομεύτηκαν τότε οι ηθικές αρχές και η αλληλεγγύη των λαών. Γιατί να πρέπει το έθνος μου να ακούει ακόμη την μοσχοβητική εκδοχή των γεγονότων. Ότι δεν υπήρξε κατοχή, ότι δεν υπήρξε το σύμφωνο Μολότοφ Ρίμπεντροπ, Γιατί ακόμη πρέπει να ακούμε τέτοια πράγματα, ότι δηλαδή αντί για κατοχή είχαμε απελευθέρωση. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν να κάνει ό,τι εξαρτάται από εκείνην για να δημιουργηθούν έρευνες για αυτά τα εγκλήματα, τις εγκληματικές ενέργειες, ώστε να καταδικαστούν δεόντως. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Φραντς Όμπενμάγερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Γερμανία και στην Σοβιετική Ένωση υπήρξε μια κατανομή σφαίρεων ε, επιρροής και οι βαλτικές χώρες βρεθήκανε στη σφαίρα επιρροής της ε, Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό οδήγησε σε μαζικές ε, εκτοπίσεις οι οποίες ακολούθησαν τη συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και ε, Σοβιετικής Ένωσης. Το 2002 το Εστονικό Κοινοβούλιο ανεκήρυξε ότι επρόκειτο για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας στην περίπτωση αυτή των εκτοπίσεων και αυτό αναγνωρίστηκε σε επίσημο επίπεδο. Η, η ενθύμηση όμως αυτών των γεγονότων είναι σημαντικό στοιχείο της ιστορίας της ε, Εστονικής, της Ανεξάρτητης Εστονίας. Στη 14η Ιουνίου λοιπόν είναι μια σημαντική στιγμή και για την Εστονία και για όλη την Ευρώπη για τα κράτη αυτά τα οποία μπόρεσαν να ξαναβρούν την ανεξαρτησία τους. Ευχαριστώ. Έχει κλείσει η συζήτηση για το θέμα αυτό και περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Λάινεν για τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. Και θα δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Γιώ Λάινεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. <clears throat> Σήμερα συζητούμε και αύριο θα ψηφίσουμε ένα